Θεωρούνται λοιπόν τα πρακτικά εγκεκριμένα. γραπτή δήλωση 71 του 2009 τον λένε ε, Μιχαήλ Τρεμόπουλου, Λίβια ε, Γιαρόκα και Τεότεγκερ για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκέντρωσε τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών σύμφωνα με το άρθρο 123 του κανονισμού και θα διαβεβαστεί αρμοδίως ε, θα συμπεριληφθεί στα κείμενα που θα εγκριθούν κατά τη διάρκεια της παρούσης συνόδου. Και θα δημοσιευθούν στα αντίστοιχα πρακτικά. Θέλει το λόγο από αυτό η κυρία Λίν. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστώ όλου του συναδέλφου που υπέγραψαν αυτή τη δήλωση περιθμών 71 για τον καρκίνο του μαστού. Όπω να ψηφίσετε περισσότεροι, πρόκειται για τον κύριο λόγο θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ηλικίε από ηλικίε 35 έω 59 ετών και θα θέλαμε να αναπτύξουμε προγράμματα διάγνωσης, έγκαιρης διάγνωσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικέ μονάδες για την ε, ε, αγωγή του καρκίνου. Πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε μια καλή δράση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βάλουμε φραγμό στις δεινές συνεπίες του καρκίνου του μαστού. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ εκείνου ε, του βουλευτέ οι οποίοι συνυπέγραψαν αυτή την ε, δήλωση. Στην Ολομέλεια τη 17η ε, Δεκεμβρίου του 2009 το Κοινοβούλιο είχε καταθέσει μια, μια, ένα αίτημα προς την νομική του επιτροπή για την, άρση της για, το, για την εξέταση ασυλίας